Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγιόγκ. Ο κύριος Λούαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ αν γέννη με τις προτάσεις του κυρίου Ντεγιόγκ, όμως θα ήθελα να κάνω και κάποιες επικρίσεις ε, και να τις συζητήσουμε. Στο σημείο ένα αναφέρθηκε στον πλουραλισμό στα ΜΜΕ και ότι οι οπτικοκουστικές υπηρεσίες έχουν το πρόβλημα της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός του, της ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος όσον αφορά τη συμπεριφορά σε κάποιες χώρες. Διαφέρει από χώρα σε χώρα η κατάσταση και κατά πολύ. Και θα πρέπει ίσως αυτό να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή όσον αφορά αυτό το θέμα. Σε κάποιες χώρες όσον αφορά το κέντρο για έρευνα για δημοσιογραφία κλπ. δεν υπάρχουν διατάξεις για περιορισμό ιδιοκτησίας. Άρα επιρροή και συγκέντρωση είναι πρόβλημα. Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ ΜΜΕ με επιχειρήσεις και με πολιτικά κόμματα. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις, ίσως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό ακριβώς ή δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Ντεγιόγκ, πράγματι υπάρχουν περίπου 7.500 φορείς ΜΜΕ που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά την επιρροή που ασκούν και την εξουσία που έχουν. Και είναι κάτι που θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό προτείνεται στο σημείο 4 του κ. Ντεγιόγκ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Έλλειψης σαφούς καθορισμού των παιδικών προγραμμάτων. Τι είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Διότι τα ΜΜΕ λένε ότι δεν επιτρέπονται διαφημίσεις εντός παιδικών προγραμμάτων. Δυστυχώς γνωρίζουμε όμως ότι 70% του χρόνου τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση μαζί με τους γονείς τους. Άρα δεν βλέπουν παιδικά προγράμματα. Και λείπει αυτός ο ορισμός, αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από την έκθεση. Και θα πρέπει να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σαφή ορισμό και να υπάρχουν σαφείς διατάξεις. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη για αυτό το ζήτημα να έχουν σαφείς διατάξεις. Και ίσως θα είχα και μία-δύο συστάσεις από την πλευρά μου και από την πλευρά του ΕΛΚ. Χρειάζεται, κατά την άποψή μου, καλύτερη κατανόηση ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών και των ενηλίκων όσον αφορά την κατανάλωση προϊόντος ΜΜΕ. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Δεν έχει γίνει μια ξεκάθαρη ανάλυση για να μπορούμε να βασιστούμε στα στοιχεία αυτά και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Πανευρωπαϊκή συγκρίσιμη μελέτη, συγκριτική μελέτη θα ήταν χρήσιμη για εκείνους που διαμορφώνουν την πολιτική στον τομέα των ΜΜΕ. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε επίπεδο κρατών θα έπρεπε να γίνει. Ίσως αυτό θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν επιτρέπετε έχω και δεύτερη πρόταση. Οι αυτορυθμιστικές προσεγγίσεις για να προσαρμοστούν συνεχείς αλλαγές του τομέα ίσως να απαιτούν περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων μεταξύ χωρών. Να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στο κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλων των εμπορευομένων, των φορέων, των επιχειρηματιών, των πολιτικών. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί πανευρωπαϊκό δίκτυο. Δίκτυο εμπειρογνωμόνων. Να συμμετέχουν εθνικοί φορείς που παίρνουν αποφάσεις και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και εκπρόσωποι των διαφόρων ε, εταιριών ΜΜΕ. Κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την ρύθμιση του ζητήματος. Ευχαριστώ κύριε Λουάν. Η κυρία Λάτφορντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ρενάτα Βέμπερ είναι η σκιώδης μας αλλά απουσιάζει αυτή τη στιγμή και με παρακάλεσε να πω ότι συμφωνεί εν γέννη με τη γνωμοδότηση, αλλά διερωτάται κατά πόσο είναι σωστό το χρονοδιάγραμμα. Η έκθεσή της, βλέπετε, για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, κινείται παραλλήλως. Νομίζω το συζητάμε το θέμα αυτό αργότερα, το απόγευμα. Μήπως Διερωτάτε, μήπως υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση του κ. Ντεγιόνγκ, φαντάζομαι ότι εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Πολιτισμού, διότι θα ήταν αρκετά χρήσιμο να δούμε και την έκθεση της Ρενάτε και να δούμε αν μπορούν να υποβληθούν συμβιβαστικέ τροπολογίες επ' αυτής και μετά να δούμε αν κάπως θα επηρεαστεί και αυτή η γνωμοδότηση, διότι η έκθεση της Ρενάτε ίσως να καλύπτει θέματα που άπτονται της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Όλα εξαρτώνται από την ευελιξία του χρονοδιαγράμματος. Θα ήμουν ευγνώμων για την άποψη του κυρίου Ντε Γιόγκ. Αυτά για την κυρία Βέμπερ. Για μένα τώρα δεν ξέρω ποιε είναι οι λεπτομέρειε της οδηγία για τις διαφημίσει στα παιδικά προγράμματα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πηγαίναμε πολύ μακριά εάν ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το δεχόμενο απαγόρευσης διαφημίσεων στα παιδικά προγράμματα, όπως προτείνεται στην παράγραφο 7. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το τι μπορεί να διαφημιστεί σε παιδικά προγράμματα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την εκμετάλλευση της αξιοπιστίας των παιδιών και της έλλειψης πείρας. Αλλά βέβαια είναι και πολύ εύπιστοι ε, και πολύ ενήλικες. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να προχωρήσουμε τόσο μακριά τόσο ώστε να απαγορευτούν οι διαφημίσεις στα παιδικά προγράμματα και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Η κυρία Αντιτσίβιτς έχει το λόγο. Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά αφού μου το δώσατε να πω δύο λόγια. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα με τα μέσα ενημέρωση σήμερα κυρίως στην Ευρώπη δεν είναι μόνο πολιτικού χαρακτήρα, αλλά και οικονομική πίεση. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ιδιοκτησία των μέσων. Και πρέπει να κάνουμε κάτι με το θέμα της ιδιοκτησίας. γιατί ε, μέσα υπάρχουν πολιτικές κατηγορίες ε, και αυτό γίνεται γιατί εκπροσωπούν ε, κάποια μυστικά συμφέροντα. Αυτό είναι προφανές. Μάλιστα, με συγχωρείτε, σας είχα στον καταλογό μου, αλλά θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ντεγιόνγκ αν θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένο από τις αντιδράσεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Λουάν. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες που εκφράσατε και αν λάβω υπόψη τις παρεμβάσεις ε, του κυρίου Λουάν και της κυρίας Λάτφορτ, κυρίως ότι αφορά τα παιδιά, θα μπορούσαμε να συντάξουμε μια νέα παράγραφο και να μας γνωστοποιηθεί ποιε είναι οι συνέπειες αυτών των διαφημίσεων επί των παιδιών και κατόπιν να ρωτήσουμε και την Κομισιόν ε, πώς ακριβώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα και για άλλα προγράμματα που δεν ε, είναι αποκλειστικά για τα παιδιά αλλά που παρακολουθούν τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν, θα πρέπει να κάνει έρευνα η Κομισιόν για τα θέματα αυτά, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογο για τα θέματα αυτά. Το θέμα τώρα της ιδιοκτησίας. Το έχω αναφέρει και πιστεύω ότι όλοι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση για το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Λόαν έκανε μια πρόταση για να συστήσουμε κάποια δίκτυα. Από την πλευρά της Κομισιόν θα ήθελα να ρωτήσω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι είναι εξαιρετική αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι υπήρχε, είναι καλό να υπάρχουν δίκτυα για να αναπτύξουμε τις βελτιστές πρακτικές. Και κατόπιν ε, μια σειρά παρατηρήσεων εκ μέρους της κυρίας Βέμπερ για το χρονοδιάγραμμα. Κοιτάξτε, επί της ουσίας, η γνωμοδότηση αυτή και η δική της έκθεση έχουν να κάνουν με το ίδιο ζήτημα. Όμως δεσμευόμαστε από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Πολιτισμού. Θα πρότεινα 15η Ιανουαρίου για τις τροπολογίες και ψηφορία 21η Ιανουαρίου. Εγώ βεβαίως ε, είμαι διαθέσιμος ε, να ακολουθήσουμε κάποιες παράλληλες διαδίκτυσεις με την έκθεση κυρία Βέμπερ, αλλά εδώ είμαι και στα χέρια της Γραμματείας και της Επιτροπής Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κομισιόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συζήτηση αφορούσε κυρίως δύο πτυχές. Ε, καταρχήν την ορθή εφαρμογή, την ίδια την εφαρμογή της οδηγίας και τις ε, πτυχές της πολιτικής. Για την ίδια την εφαρμογή η διοδηγία αναφέρεται σε συρρύθμιση και από ό,τι φαίνεται η ανησυχία των κύριων βουλευτών αφορά περισσότερο την προστασία των ανηλίκων και πώς μπορεί να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε να έχουμε κάποια κατάλληλα μέσα όπως η ρύθμιση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάλογος με τον κλάδο, με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να έχουμε αποτέλεσμα εδώ σε ό,τι αφορά την αυτορύθμιση. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πλατφόρμα και του κλάδου όπου συμμετέχουν οι σταθμοί μετάδοσης. Για το θέμα τώρα της προστασίας των ανηλίκων νομίζω ότι πρέπει να επενθυμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τους ανηλίκους υπάρχουν κανόνες στην οδηγία που αφορούν ε, τις γραμμικές και μη τις μη γραμμικές υπηρεσίες, δηλαδή την τηλεόραση, ελά και το βίντεο κατόπιν ετήματος. Ε, και εκεί λέγεται ότι επομένως ε, οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να παροτρύνουν τους ενηλίκους να αγοράσουν ή νοικιάσουν ένα προϊόν εκμεταλλευόμενοι την ευπιστία τους. Αυτό που αναφέρονται εδώ λοιπόν στο σημείο 7, δηλαδή αυτό, η πρόσκληση που ευθύνεται εδώ στα κράτη-μέλη, ήδη είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της πολιτικής, των πολιτικών. Νομίζω ότι τίθεται δύο κύρια θέματα στη συζήτηση. Έχουμε τη συγκέντρωση στα μέσα ενημέρωση αφενός και αφετέρου μία από τις πρότασεις αφορά την ευθυγράμμιση του άρθρου 21 της χάρτης και του άρθρου 6 της οδηγίας για τη συγκέντρωση των ΜΜΕ. Να υπενθυμίσω ότι συνεχίζεται η συζήτηση και στο εσωτερικό της Κομισιόν ε, και την Πρόεδρος Κρούς ζήτησε από την ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων να γνωμοδοτήσει Αναμένουμε αυτή τη γνωμοδότηση από την ομάδα, πρόεδρος της οποίας είναι ε, πρόεδρος με, σε κάποιες εβδομάδες, μια-δύο εβδομάδες και όταν ε, θα έχουμε την έκθεση αυτή θα γίνουν κάποιες προτάσεις και στην Κομισιόν αλλά και στα κρατημέλη και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευθυγράμμιση και κάποιες επισημάνσεις ε, που γίνονται στο σχέδιο κειμένου ότι δεν ε, συμπεριλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21, στο άρθρο 6 της οδηγίας, στο άρθρο 21 της χάρτας, στο άρθρο 6 της οδηγίας. Αυτή ήταν ε, η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν υιοθετήθηκε αυτό τότε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν αισθάνεται ικανοποίηση τώρα για αυτή την ε, ύστερη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορούσαμε τότε ε, να υποστηρίξουμε την πρότασή μας ε, λόγω της στάσης του συνομοθέτη. Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών προβλέπεται για τις 15 Ιανουαρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι και η ψηφοφορία προβλέπεται για την 21η Ιανουαρίου, προσωρινά. Ψηφορεί στην Επιτροπή, λοιπόν. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι οι ψηφοφορίε. Επομένω, θα πρέπει να, αναβάλουμε τη συνεδρία, να διακόψουμε τη συνεδρίαση μέχρι τι 5 και 10 προκειμένου να έλθουν όλοι οι συνάδελφοι. Για 12 λεπτά λοιπόν θα κάνουμε διάλειμμα. Συνεχίζουμε στις 5 και 10. Dear colleagues, I ask you to... Συνάδελφοι, καθίστε. Πρέπει να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. I am happy that we are so many at the vote. Χαίρομαι γιατί είναι μεγάλη προσέλευση. Καθίστε παρακαλώ. Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, αρχίζουμε την ε, ψηφοφορία. Το σχέδιο έκθεσης για το σύστημα Eurodac. Η κυρία Μακοβέ είναι η εισηγήτρια. Κυρία η θέλετε να λάβετε το λόγο πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ένας φάκελος για τον οποίο δουλέψαμε όλοι σκληρά, με διαφωνίες. Κάποια στιγμή συμφωνήσαμε επί των περισσότερων σημείων και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες και τις ομάδες για τη συνεργασία τους και ελπίζω ότι θα το τελειώσουμε το θέμα με αποδεκτή μορφή για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 61 και 62 και 63. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχέσε. Απορρίπτονται. Τροπολογία. Έλεγχος ηλεκτρονικός, αλλά ήταν σαφές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. το ΕΛΚ πέντε, τέσσερα μέλη τώρα πλέον, που είναι παραπάνω, ναι, τρεις παραπάνω, δύο παραπάνω, ένας παραπάνω, λοιπόν, ένα μέλος ακόμα είναι παραπάνω, τώρα είναι εντάξει, τώρα είναι καλά. Ψηφίζουμε. Πέρας. 39 κατά, 9 υπέρ, μία αποχή. Απορρίφθησαν λοιπόν. Τροπολογία 6 και 7 έχουν αποσυρθεί, η 64 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προτείνω να ψηφίσουμε τις 65, 66, 67, 70 και 71 μαζί, αν μπλοκ, επειδή συμφωνήθηκαν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Επί των 5 λοιπόν ψηφίζουμε μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιο είναι το πρόβλημα. 65, 66, 67, 70 και 71. Εγώ αυτές είπα να ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τώρα, οι 68 και οι 69 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αποσύρθηκε η 10 και πάμε στην 76 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Σε 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Όχι, όχι, τροπολογία 80. 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε αυτή ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 12. Περισσεύει μια ψήφος ΕΛΚ. Τώρα είναι καλά. Πέρας. 25 υπέρ, 24 κατά, δεκτή. δεν είχα την κάρτα. Κατά ψηφίζω εγώ. Και ήρθε και η πέμπτη συνάδελφος. Είναι πέμπτη κάρτα, γιατί εγώ τη δική μου δεν την έχω. Οπότε κανονικά δεν περνάει, γιατί ισοψήφισαν. Δηλαδή είναι 25 υπέρ και 25 κατά και απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν. Όταν είναι 25 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται. Ο κύριος Ταβάρες είπε στην αρχή ότι δεν έχει την κάρτα του την ηλεκτρονική και θα ψήφιζε χωρίς αυτήν. Ναι κυρία Ματιέ. Πόσους ΕΛΚ έχετε. Διότι έχουμε πολλούς ΕΛΚ που βγάλαν την ε, κάρτα τους. Έχουμε το μέγιστο αριθμό του ΕΛΚ. Me too, Αν θέλετε, μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για να τα ξεκαθαρίσουμε όλοι. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12. Πέρασε. 25 υπέρ 26 κατά. Απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13 αποσύρθηκε. Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 91. Άρχεται η ψηφοφορία. 27 υπέρ, 26 κατά δεκτή. Συγγνώμη. Αυλεψία. Η 13 έχει αποσυρθεί. 14 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έγινε δεκτή. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεκτή. 15 υπέρ κατά δύσκολο. Λοιπόν, τη 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά ε, αποχές υπέρ, υπέρ, συγγνώμη κατά πρέπει να ελέγξουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι η τροπολογία 16 αυτή που ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζεται. Πέρας. 30 υπέρ, 23 κατά. Δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 98 υπέρ, κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Περισσεύει μία ψήφος ΕΛΚ, είναι μία παραπάνω. Τώρα είναι εντάξει. Πέρας. 22 υπέρ, 32 κατά, απορρίφθηκε. 99 και 100, ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τι να κάνουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 27 κατά. Απορρίφθηκαν. 101 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχια ψηφοφορία. Πέρας. 30 υπέρ 26 κατά δεκτή. Λοιπόν, ε, ε, σε επιταχύνουμε λίγο. Η 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικά μόνο συμβιβαστικέ όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 17. Πέρας. 31 υπέρ 25 κατά δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 104 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 110, 111 και 112 ταυτόσιμες υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία 110, 111 και 112. Πέρας. 28 υπέρ, 27 κατά, δεκτές. 113 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 114 και 115 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 14 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 122 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 122 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 23 υπέρ 27 κατά 5 αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία στην 125. Έχει ένα παραπάνω το ΕΛΚ τώρα είναι εντάξει πέρα της ψηφοφορίας. 29 υπέρ 27 κατά δεκτή. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 129 είναι τμηματική. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίφθηκε. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Το δεύτερο τμήμα της 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 υπέρ 27 κατά δεκτή. Με μπερδεύετε κύριε Μωράγες με το χέρι σας. Η 130 τώρα. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία στην 132 Μία ψήφος παραπάνω στο ΕΛΚ από το κανονικό. Παρακαλώ Κάποιος πρέπει να βγάλει την κάρτα τώρα είναι καλά. Και πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 27 κατά δεκτή. 133 είναι γλωσσική, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Πάμε στην 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά έλεγχος την 137 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 29 υπέρ 27 κατά δεκτή συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 γλωσσική, δεν την ψηφίζουμε. 141 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 142 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω δεκτή. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Στην 145 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 υπέρ, 27 κατά, δεκτή. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το ιδια για τις συσχετισμοί. 147-144 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 148 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 18. Τμηματική σε πρώτο, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Πάμε τώρα στην 154 και 155 και 156 ταυτόσημες Υπέρ κατά αποχές δεκτές, 157 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα 161 Α, την 158, το πρώτο τμήμα καταπίπτει, το δεύτερο όχι. Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία όπως και πριν, αλλά για να δούμε. Πέρας. 30 υπέρ 26 κατά. Δεκτό. Και τώρα 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 με προφορική τροπολογία της κυρίας Λάτφορτ υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα θα ψηφίσουμε unblock όπως συμφώδουν οι σανιωμάδες Είναι 164, 165, 166, 167 και 169. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 167 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 100... Όχι, πάμε στην 170 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα 174-175 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 176 και 177 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 179 με προφορική τροπολογία της κυρίας Κέλλερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Πάμε στο 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στις αναφορικές σκέψεις και αιτιολογικές. σκέψεις. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 και 23 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26, 27, 29, 30 ψηφίζουμε όλες μαζί. Όχι, την 26... «26, 27, 29 και 30 λέω». «Α, όχι την 30. Καλά. Οι τρεις λοιπόν, 26, 27, 29, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 28, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τώρα, 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 15α συνδέεται με τη 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή αποσύρεται η 2 η 35 γλωσσική πάμε στην 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα οι 38, 39 και 40 να ψηφίσουμε αμπλόκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. 6α, συγγνώμη, 6α υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 2 υπέρ. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά, unblock τη 45, 47, 48, 51 και 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 55 γλωσσική, δεν την ψηφίζουμε, ψηφίζουμε την 56 υπέρ. Κατά δεν είναι σαφές. Δεν σηκώνονται καλά τα χέρια. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος, 56, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 υπέρ 27 κατά, δεκτή λοιπόν. Και ψηφίζουμε μπλοκ τις 57, 58, 59 και 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο σε τροποποιήθη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ, 11 κατά, 4 αποχές. Δεκτό. Συγχαρητήρια λοιπόν, κυρία Μακοβέη. We have no voting list. it's quite. It's quite simple. Okay. okay. Now uh, we vote on the proposal. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφασης για αύξηση του ποσοστού χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Πρόσφυγε. Εισηγητή ο κύριο Τόρβαλτ. Κύριε Τόρβαλτ, θέλετε να πείτε κάτι. Δεν διαβάζω τον μακροσκελέστατο αυτό τίτλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ εκτενώ στο θέμα. Σε πρώτερη συνεδρία συζήτησα να μην βάλετε τροπολογίε. Ήσασταν πολύ καλοί και δεν υποβάλλατε. Ήταν πολύ εύκολη δουλειά μου και σα ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τροπολογίες όσον αφορά το θέμα του Κιτόβα. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 54 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, ουδεμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Τόρβαλτς. Και έχουμε άλλη μια έκθεση του κυρίου Τόρβαλτς για το Ταμείο για τις πόλεις του Εξωτερικά Σύνορα. Δεν υπάρχουν τροπολογίες για αυτό το Ταμείο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, λοιπόν, ψηφίστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 54 ψηφίπερ. μία κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια nice Christmas holidays and I go... Λοιπόν, για τους περισσότερους σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. So uh, I will ask colleagues who want to leave the room to leave and we should continue. Παρακαλώ συνάδελφοι να αποχωρήσουμε, να αποχωρήσουν και συνεχίσουμε. Σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Τροπολογίες που υπευλήθησαν για το σχέδιο εκθέσεις χάρτης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πρότυπες διευθετήσεις σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ, την εισηγήτρια. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια καταρχάς και μετά θα έχουμε τη συζήτηση. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα πρότεινα να περιμένουμε μισό λεπτάκι για να φύγει ο κόσμος από την αίθουσα. Παρακαλώ που χωρίστε από την αίθουσα, λέει η Πρόεδρος, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ. Okay. Μπορείτε να συνεχίσετε κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τους συνάδελφους που υπέβαλαν τροπολογίες για την έκθεσή μου. Η αλήθεια είναι ότι οι τροπολογίες ευθυγνωριζόταν με τα αναμενόμενα λαμβάνοντας υπόψη τις πρώτες ανταλλαγές απόψεων επί το εγγράφου και τη δημόσια ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Γενικά, σαν σχόλιο, θα έλεγα ότι πολλές από τις ε, τροπολογίες είναι χρησιμότατες και θα εμπλουτίσουν σίγουρα την ε, έκθεση. Ήταν ευχάριστη έκπληξη διότι σε κάποια θέματα είδα ότι οι τροπολογίες ακολουθούσαν παρόμοια προσέγγιση, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα είναι αρκετά γρήγορο να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Εν γέννη, θα συμπεριλάβω πολλές τροπολογίες, θα τις υπερψηφίσω ή θα τις συμπεριλάβω στις συμβαστικές που θα προτείνω και ελπίζω το ταχύτερο δυνατόν τον Ιανουάριο να οργανωθεί μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Είναι αυτή την περίοδο του χρόνου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπω Χριστουγεννιάτικα να δουλεύει κανείς. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες, να μπω σε λεπτομέρειες, να σας πω ότι όσον αφορά την προστασία των μέσων ενημέρωσης από επιρροή, έλεγχο, απειλές, λογοκρισία, θα υποστηρίξω το περιεχόμενο των σχετικών τροπολογιών, διότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε συμβαστική τροπολογία, διαφορετικά θα ψηφιστούν οι διάφορες τροπολογίες. Όσον αφορά την παράγραφο για το μηχανισμό επιλογής διαδικασίες και για διορισμό των επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό για τη διαδικασία και για το μηχανισμό να αφήσουμε το πεδίο όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Προσωπικά θα προτιμούσα την αρχική παράγραφο της ε, έκθεσης χωρίς να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, επιλεκτικά σε κάποια κράτη-μέλη ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βέβαια όλα αυτά θα συζητηθούν ε, στις συνεδριάσεις με τους σκιώδεις εισηγητές όσον αφορά την παράγραφο για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης που είναι πυλώνας της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ποικιλομορφίας των μέσων ενημέρωσης, πρόσβαση από διάφορους φορείς ή για να εκφράζονται πολλές απόψεις, ένα ευρύ φάσμα απόψεων Ίσως μπορεί να τοποθετηθούν αυτέ οι πτυχέ σε διάφορα σημεία τη εκθέσεω, αλλά αν γέννη οι σχετικέ τροπολογίε είναι ευπρόσδεκτε. Θα έχουμε συμβαστική πρόταση για την παράγραφο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση, τα ιδιωτικά, ε, τα κρατικά και τον ρόλο που παίζουν στην κοινωνία τα μέσα ενημέρωση και των δύο τομέων, του ιδιωτικού και του δημόσιου. Στην παράγραφο 5 για την κατάχρηση των ρόλων και να επιβάλλεται έλεγχος, λογοκρισία, ε, στην ενημέρωση των πολιτών. Εκεί υπάρχουν ε, κοινέ απόψεις και όλες οι υποβληθήσει τροπολογίες θα γίνουν δεκτές. Όσον αφορά την διεκτησία των μέσων ενημέρωση, συγκέντρωση και διαχείριση και διαφάνεια, οι τροπολογίες ε, ακολουθούν παρόμοιε κατευθύνσεις, οπότε θα είναι εύκολο να συμπεριληφθούν σε συμβαστικές τροπολογίες η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων από πίεση, πρόσβαση στις πληροφορίες και ερευνητική δημοσιογραφία, όλα αυτά αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, οπότε ίσως να ενταχθούν σε διαφορετικές συμβαστικές τροπολογίες, όμως το τέλος θα αντικατοπτρίζονται στο κείμενο. Έλεγχος της κατάστασης μέσα ενημέρωσης ετησίως, Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες με τις οποίες διαφωνώ αλλά χαίρομαι διότι περισσότεροι συνάδελφοι υπεστήριξαν την πρόταση και παρέμεινε ανοιχτή η παράγραφο σχετικά με το ποιο είναι ο καλύτερος φορέας που θα διενεργεί την εποπτεία και τον έλεγχο. Δεν μπορώ να αγνοήσω την εντολή της υπηρεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι πολύ περιορισμένη. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Με χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουμε έναν οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν βρίσκονται τα χρήματα για τα μέσα ενημέρωσης. Όσο η εντολή του φορέα εξαρτάται από το Συμβούλιο πρέπει να παραμείνω να αφήσω την κατάσταση ως έχει, το κείμενο ως έχει, παρόλο που διαφωνώ. Θα συζητηθεί η ομάδα των θυμιστικών φορέων των Ευρωπαίων και πώς θα γίνει η κατανομή των εξουσιών. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις Υπάρχουν και παρόμοιες τροπολογίες περί διαφανείας, ιδιοκτησίας μέσων δημοσίων πόρων και πιστεύω ότι εύκολα θα καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά όλα αυτά. Υπάρχουν και τροπολογίες οι οποίες ακολουθούν αντίθετη προσέγγιση, δηλαδή μέχρι πού θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά τη ρύθμιση της ελευθερίας των ΜΜΕ Αυτά θα συζητηθούν στις συναντήσεις με τους σκιώδες εισηγητές και υπευλήθη σειρά τροπολογιών επί θεμάτων που δεν αφορούσαν το αρχικό κείμενο. Θα εξετάσω προσεκτικότερα τις τροπολογίες, θα τις συζητήσω το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ στον φωτοβολό των δημοσίων μέσων, τα θέματα ανταγωνισμού, χρηματοδότηση των δημοσίων ΜΜΕ, εκπαίδευση στον τομέα αυτό και διάφορα άλλα θέματα. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια και θέλω να ακούσω και ποιες είναι οι απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ρενάτα. Την κυρία Έχω στον κατάλογο με ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Ρινατέ για την εισαγωγή. Προσπαθώ να αντικαταστήσω την Κίνγκα γιατί ήταν η σκιώδη συζητριά μα, αλλά δυστυχώ έχασε την πτήση από τις ΗΠΑ και δεν μπορεί τώρα να περιβρίσκεται εδώ. Έτσι λοιπόν θα διαβιβάσω το μήνυμά της ε, εξ το τη ομάδα του Σιλστών. Η πλειονότητα των ε, τροπολογιών μας στόχευαν ζητήματα που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα όσα είπατε μόλις και παρουσιάσατε στην Επιτροπή μας. Καλούμε για περισσότερη χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε την ε, ελεύθερη έκφραση των ΜΜΕ. Πρέπει επίσης να προσαρμόσουμε τους κανονισμούς στις συγκεκριμένε ανάγκες του κάθε μέσου και υποστηρίζουμε το να θεσπιστούν κοινά πρότυπα που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία των αποπτικών έρχων και να μπορούμε να αποτρέπουμε την επιρροή από πολιτικές και οικονομικές εξουσίες. Επίσης, η πρότασή μας είναι να τροποποιηθεί οδηγία για τις υπηρεσίες ακουστικό μέσων έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι διαφανείς και αμερόληπτες και απολύτως ανεξάρτητες καλούμε για αποτελεσματικό έλεγχο της συγκέντρωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για νομικό πλαίσιο για να αποτρέψουμε τη συγκέντρωση της εξουσίας και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και ζητάμε διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης μέσω σύστασης βάσης δεδομένων έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες που αφορούν στο να συσταθούν ανεξάρτητοι ε, φορείς αυτορύθμισης και ζητούμε να υποστηριχθεί ερευνητική δημοσιογραφία κυρίως και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, ε, τονίζουμε τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων ε, και τονίζουμε ότι πρέπει οι συνθήκες εργασίας θα πρέπει να σέβονται τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εκείνη μας ανησυχία είναι ότι το κράτος και οι κρατικές εταιρείες προσπαθούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο ε, των μέσων ενημέρωσης, ανακοινώσεων των μέσων μέσω της διαφήμισης και καλούμε να υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την πολιτική πολιτική διαφήμιση ε, των κρατών. Καλούμε την Κομισιόν ε, να παρακολουθήσει αν τα δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται διαφανώ από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα δημόσια μέσα μαζική ενημέρωση. Επίση, θεωρούμε σημαντικό να εγγυηθούμε ε, ανεξάρτητα ότι θα είναι ανεξάρτητα τα δημόσια ΜΜΕ και να διασφαλίσουμε ανεξάρτητη χρηματοδότησή σας. Αυτά είναι τα μηνύματα που θα ήθελα ε, να διαβιβάσω μέσω Κίνκα και εγώ όμως έχω καταθέσει 10 περίπου τροπολογίες, ε, κυρίως προσπαθώντας να ενδυναμωθεί ο ανεξάρτητος ρόλος των ΜΜΕ και κατά της πολιτικής παρέμβασης ε, ή του εκβιασμού της δημόσιας τηλεόρασης για πολιτικούς ρόγους και επίσης στοχεύοντα και στην ε, ανάπτυξη μια ε, εναλλακτική δημόσια τηλεόραση, όπως έγινε πρόσφατα στη Σλοβενία, στη χώρα μου. οι τροπολογίε ε, στοχεύουν στο να τιμωρηθούν όλοι όσοι επιτίθενται στου δημοσιογράφου. Πολύ συχνά έχουμε κάποιε διαδικασίε, αλλά δεν ολοκληρώνονται. Δεν έχουμε λοιπόν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ε, κατά όσων ε, εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Αναμένω λοιπόν ότι η συγκήτρια θα συμφωνήσει με τις τροπολογίες μας, καθώς όλες θέλουν να ενδυναμώσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Όλες οι τροπολογίες επικεντρώνονται στον κώδικα δεντολογίας, ε, στη διαφάνεια του διευθυντικού καθεστώτος, των ΜΜΕ. Υπάρχει και μια πρόταση σε σχέση με μια Ένωση Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Αν δούμε το ψήφισμα αυτό, έχω την εντύπωση ότι έχουμε σχεδόν ε, τα τέλεια μέσα μαζικής ενημέρωση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σταβάρης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη Ρενάτε Βέμπερ. Είναι, ήταν έξοχη συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει στην έκθεση να ακολουθήσουμε τον προβληματισμό που εκφράζουν οι πολίτες μας. Δηλαδή η ελευθερία των μέσων κινδυνεύει λόγω της οικονομικής καταστάσεως που συνεχώς αλλάζει και επιδεινούνται τάχιστα, οπότε πρέπει να κάνει κάτι ένωση γι' αυτό, διότι δεν είναι πλέον τοπικά τα μέσα, όλα τα ΜΜΕ έχουν στο σελίδες, έχουν υπερεθνική διεθνή εμβέλεια, οπότε θα πρέπει να δει και αυτή την επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε δημοκρατία, πληρολισμό και σεβασμό μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 στη συνθήκη και θα πρέπει να εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα. Και η δημοκρατία και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Ε, ήταν αρχές που εφαρμόζονται το 18ο και 19ο αιώνα. Αυτή είναι η θεωρητική πτυχή. Η πρακτική είναι ότι αλλάζει πολύ γρήγορα η κατάσταση. Έχουμε τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζει το επιχειρηματικό μοντέλο σημαντικού τομέα των μέσων ενημέρωσης και θα πρέπει να βοηθήσουν οι δημόσιοι φορείς στη μετάβαση και την αλλαγή που απαιτείται να μην διασωθούν θνήσκουσες επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια για να γίνει σωστή μετάβαση όλες αυτές τι ιδέες πρέπει να τις μεταφράσουμε σε τροπολογίες. Χαίρομαι ότι η Ρενάτε θεωρεί ότι οι υποβληθεί τροπολογίες ήταν καλές και το θέμα των προσωρινών ε, της ανασφάλειας της εργασίας στην δημοσιογραφία, διότι ε, ένας δημοσιογράφος που δεν αισθάνεται ασφαλής δεν πάει να κάνει καλά τη δουλειά του, δεν αισθάνεται ασφαλής όσον αφορά τη θέση του. Έχουμε την Ειδική Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα, Διαφθορά και Ξέπλυμα Χρήματος που συζητά το θέμα προστασίας της ερευνητικής δημοσιογραφίας για να αποφύγουμε στο μέλλον διάφορα οικονομικά εγκλήματα που θα υπάρχουν. Αν δεν είναι εξάρτητη δημοσιογραφία κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και αυτά θα φανούν στο μέλλον και θα έχουμε νέα κρίση στο μέλλον. Τεχνολογική αλλαγή λοιπόν και η ανασφάλεια όσον αφορά τις θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων. Γι' αυτό θέλουμε να κάνει μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μελετήσει τι συνέπειες έχουν οι αλλαγές και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Μία ανάλυση των φαινομένων αυτών είναι κάτι επίμαχο, τα ε, αφήσαμε στο επίπεδο μελέτης, που είναι το σωστό επίπεδο σε αυτή τη φάση, για τα φαινόμενα. Τα άλλα σημεία σωστά τα περιέγραψε η ίδια Ρενάτα. Οπότε περιμένω μελλοντικέ επαφέ απέσυνδεδών και συνεργασία. Ευχαριστώ ο κύριο Ιόγκ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και πάλι, νομίζω πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. είναι οι προτεραιότητες κατ' εμέ. Πρώτον, οι ιδιοκτησιακές σχέσεις και θέματα συγκέντρωσης των μέσων. Δεύτερον, ε, ο σημαντικός ρόλος των ε, δημοσίων ΜΜΕ και τρίτον η ενθάρρυνση της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη και σε σχέση με την Ειδική Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα έχουμε το ίδιο θέμα. Είναι πολύ σημαντική εκεί η ερευνητική δημοσιογραφία. Τέλος, μετά την, ε, τις 11 Σεπτεμβρίου πρέπει να ανοίξουμε προς τους πολίτες ε, να έχουμε δημόσια ενημέρωση, ε, οι κυβερνήσεις δηλαδή για τους πολίτες και είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό. Αυτές είναι οι βασικές τέσσερις προτεραιότητες, αλλά δεν άκουσα τίποτε στην παρέμβαση της Ρενάτε Βέμπερ που να λέει κάτι διαφορετικό. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον την συνάντηση των σκιωδών και συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας. Και τώρα η Ρενάτε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις. Ε, τώρα είναι θεωρητικό ερώτημα. Αν συμφωνούμε τόσο πολύ αυτό συμβαίνει γιατί δεν πιάσαμε τα πιο ευαίσθητα θέματα ή όντως επειδή αντιληφθήκαμε μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων ε, πάνω στα προβλήματα γιατι ειναι η ελευθερία των ΜΜΕ ότι πράγματι πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτό ομονοούμε. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση όλοι δηλαδή. Εγώ έχω πιστεί ότι τώρα είναι πια η ώρα να είμαστε πιο ξεκάθαροι, πιο αυστηροί, να λειτουργήσουμε σε βάση ρυθμιστική όταν μιλάμε για τα προβλήματα των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας. Και είμαι βεβαία ότι αρκετά πολύ εύκολα θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Επίσης σημείωσα και από τις τροπολογίες και ακούγοντας σήμερα και τους συναδέλφους βλέπω ότι υπάρχει αυτό το στεναρό αίτημα να προωθήσουμε και να έχουμε ε, στιβαρό, στιβαρή ε, ερευνητική δημοσιογραφία και θα πρέπει να υποστηριχθεί και από δημόσια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διατεθούν και τέτοιες πιστώσεις από μας. Δεν ξέρω ε, αν συμφωνείτε όλοι με αυτή την προσέγγιση. Θα το συμπεριλάβω αυτό το σημείο στην έκθεση. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω, ε, μόνο τις ευχές μου ε, θα προσθέσω για τις γιορτές και θα ειδωθούμε πάλι του χρόνου. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή στις 21 και 22 Ιανουαρίου. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για τις εορτές των Χριστουγέννων. Τώρα αύριο θα συνεχίσουμε ε, όμως εμείς θα αρχίσουμε στις 9 το πρωί με τα συμπεράσματα των επιτευμάτων της Κυπριακής Προεδρίας και το απόγευμα θα έρθει και η κυρία Ρέντινγκ στις 3 η ώρα. Οπότε τα μέλη που μπορούν παρακαλώ να έρθουν. Ευχαριστώ. Τώρα διακόπτεται η σημερινή συνεδρίαση.